Bonsoir à toutes et à tous. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Βρυξέλλας και θα έχουμε άμεση μετάδοση, απευθεία μετάδοση αυτής της συζήτησης για ε, τι κοινωνικέ πτυχέ τη οικονομική κρίση. Είχαμε αυτή τη ε, συζήτηση που θα μεταδοθεί και στο Βουκουρέστι και εκεί που έχουμε καλέσει τώρα τον, τον ε, κύριο Μανσίν, τον Επίτροπο Μπαρό, τον Φιλίπ Ντεμπίκ που είναι ο, ο διευθυντής ε, του φορέα που αντιπροσωπεί του τους επιχειρηματίες στην Ευρώπη, τον κύριο Χόφμαν, επίσης από τη Συνομοσπονδία των Συνδικάτων και, και ε, να σα αρχίσουμε πρώτα-πρώτα με τον κύριο Μαντσίν, αν μπορείτε πέστε μας δύο λόγια όσον αφορά αυτή ε, την τελευταία φάση των εκλογών. Όσον αφορά την αποχή, είχαμε πει ότι θα υπάρξει εντυπωσιακή διαφορά, εντυπωσιακή πτώση, τελικά αυτό δεν έγινε. Αυτό συνέβη μόνο μέχρι σε ένα συγκεκριμένο βαθμό σε ορισμένε χώρε. Όμω, σε κάποιε μεγάλε χώρε όπω τη Γερμανία, το πιο πρόσφατε διαπιστώσει αφορούν ένα 0,5% διαφορά μεταξύ των προηγούμενων ευρωεκλογών και των φετινών. Σε ορισμένε εκλογέ δε διαπιστώσαμε αύξησε τις προσέλευσεις. Φερρυπίν, στη Βουλγαρία εντυπωσιακή αύξησε. Στην Λετωνία. Σε κάποιες χώρες όπου ε, ήταν πολύ έντονος ο προβληματισμός των ε, ψηφόρων ακόμα και στην Ιρλανδία. Κατέβηκαν να ψηφίσουν οι πιο πολλοί από ότι ποτέ. Περί το 61% κατέβηκαν να ψηφίσουν. Και τώρα. Κύριε Μπαρό. Καλησπέρα σας. Κατά τη γνώμη σας, η εσωτερική αγορά είναι δυνατόν να προχωρήσει χωρίς να υπάρχει κοινωνική Ευρώπη, να, τον, να την διαχειριστούμε. Ο, ναι, θα πρέπει να συγκεράσουμε από τη μία μεριά την ε, δυναμική ιστορική αγορά με τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί, να συγκεραστεί με την κοινωνική πολιτική. Αυτό πρέπει να γίνει από το Κοινωνικό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να συγκεράσει αυτό που σημαίνει δυναμισμός ιστορικής αγοράς ε, να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την απελευθέρωση όσον αφορά τη ρύθμιση του ανταγωνισμού, αλλά επίση θα πρέπει να δοθεί και αυτή η κοινωνική πτυχή. Κατά τη γνώμη μου, απαιτεί αυτό ε, το να επιστατεύσουμε περισσότερου πόρου, απλούστευση των διαδικασιών, τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Δεν θα πρέπει να αποστερηθούμε αυτών των ανθρωπινών πόρων. Για αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προσέξουμε το πώς θα διασώσουμε τους μισθωτούς. Ναι, αλλά πέστε μας, γιατί δεν τα κατάφεραν οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα. Και δεν μιλώ για τους πολιτικούς, μιλώ και για τους συνδικαλιστές η συνομοσπονδία μας ανέκαθεν τόνιζε την κοινωνική πτυχή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και μέχρι ενός βαθμού είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό το ότι είχαμε αυτή τη συμμετοχή στις ε, εκλογές. Ακόμα έχουμε μεγάλη εποχή, αλλά θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Θα πρέπει την επόμενη πενταετία, επομένω να έχουμε ένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έχουμε μπροστά μας μια τρομερή κρίση η οποία θα οδηγήσει σε τρομερές συντάσεις στην αγορά εργασίας. Αυτέ θα πρέπει να υπεργεράσουμε και η Ευρώπη θα πρέπει τώρα να αποδείξει ότι θα είναι πετυχημένη, θα μπορέσει να δρώσει την ενιαία αγορά και το κοινό νόμισμα μόνο εάν προσέξει αυτή την κοινωνική πτυχή. Όλοι χρειαζόμαστε μια αυθεντική κοινωνική ολοκλήρωση. Κύριε Ντεμπούκ, υπέρ, η μόνο δεν είναι όταν υπάρχει μια τέτοια ισχυρή κοινωνική πτυχή. Υπέρ των γενικών εταιριών δεν είναι, ναι, είναι για το συμφέρον της Ευρώπης του να έχει μια ισχυρή εσωτερική αγορά, κάτι το οποίο στο παρελθόν το καταφέραμε. Και είχαμε ένα σωρό θετικές συνέπειες. Εκατομμύρια θεσμοργασίες δημιουργήθηκαν ως εκ τούτου. Κοινωνική Ευρώπη όμως δεν σημαίνει πόσους νόμους και κανόνες θεσπίζει κανείς και πόσες συμβάσεις συνάπτει κανείς. Συγγνώμη που θα πρέπει να σας ε, διακόψω διότι θα πρέπει τώρα να δούμε τι γίνεται στη Ρουμανία. Σε απευθεία σύνδεση με τον συνάδελφο Λούκα Νικολέσκο. Οπότε θα δούμε ε, τι ακριβώς, πώς έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις στην Ρουμανία. Λούκα, βρίσκεσαι στο στούντιο της ε, Ρουμανικής Τηλεόρασης. Καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά τις, ε, τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρουμανία. Καλησπέρα σας. Οι τελευταίες τάσεις μόλις έφτασαν τα δύο μεγάλα κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό Αριστερό Κόμμα και το Ελεύθερο ε, Δημοκρατικό, το δεξί, ε, είναι διαφορά στήθος με στήθος, 30% περίπου και υπάρχει και ένα τρίτο κόμμα, το Φιλελεύθερο με 16% αλλά η μεγάλη είδηση, γιατί είναι τάσεις βέβαια, είναι ε, η είσοδος της ακροδεξιάς με 7% που ε, μάλλον θα επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου είχε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Κατά την άποψή σας κύριε Νικουλέσκου, υπήρξε αρνητική επίπτωση της οικονομικής κρίσης επί των επιλογών των ε, Ρουμάνων πολιτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αύξηση της άκρας δεξιάς. Συνήθως αυτό συνδέεται με μια κοινωνική δυσφορία. Βεβαίως, διότι η άκρα δεξιά πραγματικά έκανε εκστρατεία ε, σε αυτό, στην κοινωνική ε, δυσφορία των Ρουμάνων και την οικονομική κρίση. Βέβαια το θέμα αυτό δεν το συζήτησαν πάρα πολύ, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα που σας προανέφερα μετέχουν και τα δύο στον κυβερνητικό συνασπισμό. Αριστερά-δεξιά συγκυβερνούν. Επίση, θα πρέπει κανεί να γνωρίζει ότι η οικονομική κρίση μπορεί με να είναι παρούσα, αλλά δεν κυριαρχεί τόσο πολύ όπω σε άλλε χώρε. Για παράδειγμα, η ανεργία στη Ρουμανία είναι μόλι 5% σε σχέση με την Ισπανία, α πούμε, ακόμα πολύ περιορισμένη. Επιπλέον, Υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν και πολύ καλά. Η Dacia Φερρυπίν που ε, κατασκευάζει εδώ το μοντέλο Logan. Ε, αυξάνεται η παραγωγή τη όλο και περισσότερο από τις αρχές του έτου, γιατί υπάρχει ε, στη Γαλλία και στη Γερμανία πριν απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων. Οπότε τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη Ρουμανία ε, είναι ευπόλυτα παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Νικολέσκου. Κύριε Ντεμπούκ. Λοιπόν, το σύστημα προστατευτισμού ε, στην αυτοκινητομηχανία ισχύει και στις άλλες χώρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα που θα πρέπει να εξάγουμε. Μιλούμε για την ενιαία εσωτερική αγορά εδώ και γνωρίζουμε ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο για σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά αν κάποιος λαμβάνει μέτρα σε μια χώρα εις βάρος μιας άλλης, αυτό είναι αρνητικό για όλους. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι κομβικό ζήτημα η εσωτερική αγορά, όχι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Και με τον συνάδελφο μου, τον Ράινα Χόφμαν, προσπαθήσαμε να ε, καταλήξουμε σε συμφωνίε. Ποτέ όμω δεν θα καταφέρουμε να έχουμε συλλογικέ διαπραγματεύσει για του μισθού πανευρωπαϊκά. Πώ μπορεί αυτό να ε, συνδυαστεί, α πούμε, Ρουμανία με Γερμανία. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε κοινού μισθού. Θα πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη αυτά τα νέα να φτάσουν ε, στο επίπεδο των παλιών. Κύριε Επίτροπε, πώς μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα προβλήματα, αυτές οι διαφορές, η ψαλίδα η τεράστια που υπάρχει. Ενδεχομένω αυτό μπορεί να καταστρέψει την εσωτερική αγορά. Είναι τεράστιο χάσμα αυτό, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, λέει ο Επίτροπος κύριο Μπαρό. Το πρώτο μας μέλημα είναι η απασχόληση. Και εκεί η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει το ρόλο που τη αναλογεί. Άκουσα τον κύριο Ντεμπιού, κατανοώ τα όσα λέγει ε, προ του μισθού κάθε κράτο μέλο έχει ακόμα αρμοδιότητες αναμφισβήτητες. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση οφείλουν να βοηθήσουν και πραγματικά να δώσουν κίνητρα στα κράτη-μέλη να ε, διαφυλάξουν, να διατηρήσουν την απασχόληση με μερική ενεργεία όπου χρειάζεται, με επιμόρφωση των εργαζομένων για νέα επαγγέλματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει τον ανθρώπινο πλούτο της. Γιατί όμως τα συνδικάτα έδρασαν σε εθνικό μόνο επίπεδο. Καθόλου ε, ο εκπρόσωπος των συνδικάτων τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνομοσπονδία μας λειτουργεί από το 1973 που ιδρύθηκε και έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο για να υπάρξει μια κοινωνική διαμόρφωση των ε, διεκδικησιών. και ε, Άλλε φορέ ε, επιτυχάνουμε, ε, άλλε φορέ όχι. Αυτό που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει είναι το εξή. Για παράδειγμα, αν ο κύριο Ντεπούκ υποστηρίζει και υπογραμμίζει ότι δημιουργούμε νέε θέσει απασχόληση, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανισότητε στην Ευρώπη. Πόσε από αυτέ τι νέε θέσει απασχόληση είναι επισφαλεί, άραγε. Τι μπορούμε να κάνουμε συμπληρωματικά με τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο Εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, χρειάζεται μια γνήσια ε, κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη. Κύριε Μαντσίν, είδατε κάποιες δημοσκοπήσεις. Ε, εσείς τι πιστεύετε. Θεωρείτε ότι υπάρχει ενιαία αντίληψη στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες μέλη, ε, ως προς την κοινωνική Ευρώπη. Απάντησε, κύριο Στεμπιούκ. Κοιτάξτε, Το θέμα είναι αν οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη ως τη λύση των προβλημάτων τους, την άμεση λύση για τα όσα τους απασχολούν. Εκεί είναι το μεγάλο χάσμα. Όταν τους ρωτάς σε ποιο επίπεδο θεωρείς ότι θα λυθούν τα προβλήματά σου, μόλις το 9% απαντά το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το υπόλοιπο περίπου ε, μοιράζεται ανάμεσα στην εθνική κυβέρνηση περίπου ένα 50% και ένα 38% σε περιφερειακές κυβερνήσεις. Δηλαδή θεωρούν την Ευρώπη κάτι πολύ μακρινό από την καθημερινή του ζωή. Ας πούμε. Αν ρωτήσαμε τι γίνεται με την οικονομική ε, κρίση, μπορεί να λυθεί σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό ή σε, κρατικό και λένε όχι, όχι. Ε, θεωρούν ότι ε, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και αφορά και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουν μεγάλες μεν προσδοκίες από την Ευρώπη, αλλά δεν το βλέπουν πάντα ως λύση το ευρωπαϊκό επίπεδο και κάτι πραγματικά είναι πραγματικό χάσμα αυτό στην Ευρώπη. Είναι πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες ε, στη δική τους παρουσία και στην καθημερινή τους ζωή. Δηλαδή πόσο επηρεάζει η Ευρώπη την καθημερινή σου ζωή. Στις κάτω χώρες ας πούμε ένα 5% το πιστεύει. Ενώ ε, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Βλέπετε εκεί η διαίρεση δεν πάει παλιά κράτη-μέλη, νέα κράτη-μέλη, ούτε γεωγραφικά. Ε, το θέμα είναι λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι επιτράει η Ευρώπη στην καθημερινή του ζωή. Α πάμε στο Βουκουρέστι. Συνδεόμαστε με το Βουκουρέστι και καλωσορίζουμε τον Επίτροπο κύριο Όρμπαν. Καλησπέρα σα κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα. Εσεί τι πιστεύετε, πώ ψήφισαν οι Ρουμάνοι και είναι απογοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, λέει ο κύριος Επίτροπος. Μεγάλη είναι η πλειοψηφία των ε, Ρουμάνων πολιτών υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονό ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ υψηλή, σχετικά χαμηλότερη από τι ε, προηγούμενε εκλογέ του 2007. Πάντως, μπορώ να σα πω ότι βλέπουμε ξεκάθαρα πλειοψηφία των Ρουμάνων υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε τελικά να πείσει τους Ρουμάνους πολίτες. Διότι ανεξάρτητα από την έκβαση του αποτελέσματος, ε, ε, είναι εύγλωτα τα αποτελέσματα αυτά. Δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντά ο κ. Σόρμπαν. Νομίζω θα πρέπει να συγκρίνουμε τη συμμετοχή στι εκλογέ με τη συμμετοχή στι πρόσφατε βουλευτικέ εκλογέ, που ήταν κάτω από 40%. Δηλαδή, είναι πραγματικά η συμπεριφορά και η στάση του πληθυσμού τη Ρουμανία ε, ω προ το δικαίωμα ψήφου που έχουν. Και επίση δεν έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλε συζητήσει, τηλεμαχίε. Ε, ε, δημόσια αντιπαράθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρξε έτσι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε ε, για ε, τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Επίτροπε, κύριε Βαρό, εσείς θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει κάνει και λάθη στη διαχείριση της κρίσης γύρω στο Σεπτέμβριο, ας πούμε. Μήπως δεν κατάφερε να ε, παρουσιάσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα ανάκαμψης οικονομίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, ο κύριος Μπαρό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι γεγονός ότι για την κρίση νομίζω προσέκρουσε σε κάποια πάρα πολύ εθνικά ανακλαστικά από πλευράς κυβερνήσεων. Και σε μια πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε το σχέδιο υποστήριξης ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης να είναι ευρωπαϊκό. Πάντως έπαιξε ένα ρόλο συντονιστικό από την αρχή και είχε πραγματικά και ένα αντανακλαστικό να εγγυηθεί τις τραπεζικές καταθέσεις των μεμονωμένων πολιτών. Ε, ε, έλαβε τα μέτρα που έπρεπε για να μην κατακαιρματιστεί η προσπάθεια στην Ευρώπη. Είναι γεγονός όμως ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγεί ακόμα καλύτερα ε, το τι πράττει για να ρυθμίζει τις χρηματαγορές και να υποστηρίζει την οικονομία. Για να γίνει όμως αυτό σίγουρα θα χρειάζεται πιο φιλόδοξος και προπολογισμό. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα συμφωνούν. Η παρούσα επιτροπή του κυρίου Μπαρόζο έκανε το καθήκον της. Νομίζω ότι η επιτροπή αυτή θα μπορούσε να ε, είχε αποδειχθεί περισσότερο φιλόδοξο, φιλόδοξη, πολύ περισσότερο από ό,τι εφάνηκε τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράδειγμα, είδαμε τι έγινε με τι αποφάσει του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είναι πάρα πολύ ισχυρά τα μηνύματα που στέλνουν και λάθο μηνύματα στου πολίτε. ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, θέτει τι οικονομικέ ελευθερίε ε, υπεράνω των ε, βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων. Χρειάζεται διευκρίνηση και νομίζω ότι ε, είχε την ευκαιρία και θα έπρεπε να το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα προέχουν είναι σημαντικό για τον κόσμο αυτό. Οι πολίτε πιστεύουν στην Ευρώπη, αλλά έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη αυτή. Και ειδικά με την κρίση αυτή που ζούμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο φιλόδοξοι. Η οδηγία για το χρόνο εργασία δεν ήταν πιστική, αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ήρθε τώρα μετά τι αποφάσει του δικαστηρίου και προσπάθησε να ερμηνεύσει ε, τι αποφάσει ε, και τι οδηγίε με τρόπο παράδεκτο και στέλνει και λάθο μηνύματα. Ναι, αλλά ας πούμε όταν έχουμε την ε, συγκεκριμένη περίπτωση της αυτοκινητομηχανίας Opel, αλλά και άλλων, στη Γαλλία, την Ιταλία και παντού στην Ευρώπη. Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και τα συνδικάτα και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιθυμούν περισσότερη Ευρώπη. Βεβαίως και επιθυμούν. Ή μήπω υπάρχει ένα είδος οικονομικού εθνικισμού και εκεί. Εγώ είμαι σε πολύ στενή επαφή με τους συναδέλφους της Όπελ, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιχείρησης και πραγματικά προσπαθούν να βρουν ευρωπαϊκές λύσεις. Όχι μόνο μια λύση για τους εργαζόμενους στην Όπελ της Γερμανίας. Αυτό όμως που μας χρειάζεται είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αυτοκινητοβιομηχανία γενικώ. Δεν έχει νόημα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έχει κάθε χώρα ξεχωριστά. Χρειάζεται ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική παντού. Εσεί νομίζετε ότι υπάρχει πραγματική βούληση από πλευρά ευρωπαϊκών συνδικάτων για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα κοινωνικά προβλήματα. Να ρωτήσετε τον κύριο Χόφμαν, λέει ο εκπρόσωπο της εργοδοσίας. Ναι, θα επανέλθω όμω. να απαντήσω λίγο σε αυτό που ανέφερε ο επίτροπο, γιατί η ερώτησή σα ήταν ε, ουσιαστικότατη. Λειτουργήσαν σωστά τα θεσμικά όργανα όταν ξέσπασε η κρίση. Εγώ απαντώ ε, ναι, διότι οι πρώτοι που επενέβησαν με τρόπο ριζικό και θετικό ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, στη συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια τη Γαλλική Προεδρία με μεγάλη πυγμή και ισχύ για να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν όλου του ενεχόμενου που είχαν λόγο ή είχαν μέσα να δράσουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα δεν ξέρει ότι καμιά φορά εκφράζω και επικρίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να είμαστε όμω άδικοι απέναντί τη. Γιατί προσπάθησε να συγκεντρώσει όλου του ενδιαφερόμενου και κατάφερε να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εθνικά σχέδια. Και τα 5 δισεκατομμυριάκια που είναι στα γόνα στον ωκεανό χρειάστηκαν μήνες για να εκταμιευθούν και για να ε, συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στα θεσμικά όργανα και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι πάντα πρόκειται για συνδυασμό μεταξύ των όσων γίνονται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και το μέγα δίδαγμα από την κρίση αυτή νομίζω είναι το εξής. Και θα πρέπει να το αναλάβει το νέο κοινοβούλιο που μόλις εκλέγεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα νέα όργανα, είναι πραγματικά να εξηγήσει στους πάντες ότι μόνο με ευρωπαϊκή λύση θα βγούμε από την κρίση αυτή. Αυτό είναι το μέγα δίδαγμα και μήνυμα. Κύριε Μάντσιν, τι αναμένουν οι Ευρωπαίοι από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ως τα κοινωνικά και τα οικονομικά θέματα. Περιμένουν πράγματα όχι πάρα πολύ αφηρημένα. Τα πρώτα αποτελέσματα καμιά φορά μπορεί να φαίνονται και συγκλονιστικά. Πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30% και 36% στην Αυστρία πηγαίνει σε κόμματα ευρωσκεπτιστικά. 18% παίρνει ο κύριος Χάντς Πέτερ Μάρτιν, που είναι σαφής επικριτής ε, της Ευρώπης και ορισμένων ευρωβουλευτών. Αντίστοιχα συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, από τη μια οι πολίτες θέλουν να έχουν και προσωπικές σχέσεις και απαιτούν και ε, ακαιρεότητα και όχι πολλά γενικά και αφηρημένα. Τώρα, για το κατά πόσο επηρεάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη ζωή τους ε, υπάρχει μεγάλη αμφιθυμία. Θέλουν βέβαια κάποιος να κάνει κάτι από την άλλη όμως υπάρχουν και πολύ διαφορετικοί πολιτικοί πολιτισμοί ανά την Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες επιστέφονται περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λιγότερο την κυβέρνησή τους. Γιατί θεωρούν ότι είναι ο έξωθεν έλεγχος της ίδιας της κυβέρνησης. Πάντως τελικά λιγότερο από το 15% των ε, κομμάτων Ε, έχουν το αποτέλεσμα που περίμενε. Κύριε Επίτροπε, χωρίς μεγαλύτερη χρηματοδότηση όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι γίνεται λοιπόν με τον κοινοτικό προπολογισμό. Δεν θεωρείτε ότι είναι κάπως περιορισμένος. Κοιτάξτε, εμεί πιστεύουμε πάρα πολύ στη συμμαχία Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είδαμε, α πούμε, για του οργανισμού βαθμονόμηση που εν μέρει οφείλονται για την κρίση. Έγινε πολύ καλή συνεργασία. Η πρωτοβουλία και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο πάρα πολύ δραστήριο και αποτελεσματικό. Τώρα, είναι γεγονός ότι σήμερα δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη. Και ξέρω γιατί μιλώ, γιατί ήμουν αρμόδιος για τις υποδομές. Ε, χρειάζεται πραγματικά να έχει αυτόνομη δυνατότητα δανειοδότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει αρκετούς ε, ιδίους πόρους. Άρα δηλαδή αύξηση του προπολογισμού τα δημοσιογράφηση. Ναι, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε κάνει καλή δουλειά. Α μην λησμονούμε την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Εσεί τι λέτε για τον προπολογισμό, θα πρέπει να αυξηθεί ο εκπρόσωπο του Συνδικάτου. Ναι, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, άρα και μεγαλύτερο κοινοτικό προπολογισμό. Περισσότερε επενδύσει από τα διορθωτικά ταμεία στην καινοτομία. Χρειάζεται επίση ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και όλος ο προϋπολογισμός σήμερα είναι το 1% του ε, ΑΕΠ. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ε, συμμετοχή και ένας, ε, ε, ε, ένας ευρωπαϊκός φόρος. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί, δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Αν αναλύσουμε τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών και δούμε πόσο χαμηλή ήταν η συμμετοχή, το θέμα δεν είναι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αντιδρά έτσι και κατά των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπου τι αποβάσεις όμως τι παίρνουν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Κύριε Ντεμπούκ, δεν νομίζετε ότι ε, περισσότερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημάνουν και μεγαλύτερε δαπάνε. Βέβαια, όταν έχει περισσότερα χρήματα, ε, σημαίνει μεγαλύτερε δαπάνε. Άμα δίνει λεφτά σε ένα πολιτικό, θα τα δαπανίσει. Τι θα τα κάνει. Το θέμα όμω είναι και το ζήτημα ότι ποιο θα ε, κάνει αυτέ τι μεταφορέ των πιστώσεων. Γιατί αν αυξηθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνοντα του φόρου, δεν είναι αυτή η λύση βεβαίω, έτσι. Εκεί είναι το στοιχείο κλειδί τη μεταφορά των πόρων. Και, και δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο μεταφορά πόρων, χρημάτων δηλαδή, αλλά και χώρη εξουσιών. Και αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Αλλά μια που με ρωτήσετε για τα συνδικάτα, εμείς είμαστε ανοιχτοί στον κοινωνικό διάλογο και πρόθυμοι πάντα. Γνωρίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα είναι συστήματα κλειδιά και σε περίοδο κρίσης. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε επίση επίγνωση ότι απομένουν πολλά να γίνουν σε εθνικό επίπεδο και δεν είναι ότι δεν θέλουμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο και εκεί πρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όποιο θέλετε, αλλά πραγματικά με αγωνία ε, ενδιαφερόμαστε για το ποιο είναι το σωστό επίπεδο να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μισό λεπτό έχετε κύριε Μαντσί να μας πείτε τι περιμένουν οι πολίτες από το μεγαλύτερο προπολογισμό και την περισσότερη Ευρώπη. Ε, είναι θέμα πάρα πολύ επίμαχο. «80-90% για τα κοινωνικά θα πούνε ναι, αλλά το θέμα είναι πώς ρωτάς. Άμα το ρωτήσεις και θες να βάλεις πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη με καλύτερους φόρους, 80% θα σου πει όχι. Μα είναι επενδύσεις, λέει ο κύριος Μπαρό. Επενδύσεις. Περί αυτού πρόκειται. Το θέμα δεν είναι η Ευρώπη να γίνει σπάταλη στη λειτουργία της, στις λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις. Και ξέρω γιατί μιλώ, ξέρω ότι είναι τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα που για σήμερα πραγματικά θα ήταν ενδιαφέρον να επιταχύνουμε λίγο τη λειτουργία και να δώσουμε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους σας ε, για τη συμμετοχή στη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε και το Βουκουρέστι. Λιόν, σε εσά ο λόγος τώρα.